η πρόεδρος Ουλφ Σκόγκ. Αρχίζουμε την ε, συνεδρίασή μας. Την επαναλαμβάνουμε μάλλον. Αφού έχουμε τους προσκεκλημένους από τους οργανισμούς, και μάλιστα από τότε που αρχίσαμε, αναλάβαμε τα καθηκοντά μας ως νέοι ευρωβουλευτές, δηλαδή με την επανέναξη των εργασιών του Κοινοβουλίου. Τώρα έχουμε τους οργανισμούς κοντά μας, οι οποίοι θα αναπτύξουν τα πεπραγμένα τους ατομικώς, σχετικά με το τι έχουν κάνει και ποια είναι τα σχέδιά τους για το επόμενο χρόνο ή τα επόμενα χρόνια. Κάθονται κάτω στα καθέσματά τους, στην αίθουσα, οι διευθυντέ και διευθύντριε και θα κάνουν μια σύντομη παρουσίαση και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα αρχίσω λοιπόν με τον κύριο Καλέχα που είναι Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ ορίστε στα αγγλικά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες και αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί φέρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντύτερα στις ανάγκες των πολιτών. Η παρουσία των οργανισμών στις διάφορες χώρες μέλη συμβολίζει επίσης το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει στους πολίτες της και χρειάζεται την έμπνευση από αυτούς που σε αυτήν στηρίζονται και οι δραστηριότητες των οργανισμών. Ιδρυθήκαμε το 1975 και αυτό μας κάνει μαζί με τον Eurofound τον παλαιότερο οργανισμό. Είχαμε λοιπόν ιδρυθεί τότε στο διαιρεμένο Βερολίνο και το 1995 μετακομίσαμε από το ενωμένο πια Βερολίνο και μεταβήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά τα χρόνια, 40 χρόνια, η προστιθέμενη αξία που δίνουμε είναι για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση. 40 χρόνια, όπως είπα, πολλές αλλαγές και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα που περιλαμβάνουν και, τις, και τους στόχους της Ένωσης για ανάπτυξη και απασχόληση απαιτούν τώρα πια νέες προσεγγίσεις για τη μάθηση για να βρει κανείς δουλειά. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα διαρκώς ανανεούμενο όραμα για το ποια θα είναι η μορφή των νέων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για το λόγο αυτό ο ΣΕΝΤΕΦΟΠ έχει επιλέξει ένα μότο, ένα σύνθημα ότι όλα οδηγούν σε νέους δρόμους. Οι παλιοί δρόμοι στους καινούριου δρόμους. Οι παλιοί πρέπει να γίνουν καινούργοι, δηλαδή μονοπάτια, προσεγγίσεις, ευκαιρίες για σταδιοδρομίες και δουλειά. Οι παλιοί δρόμοι των ε, εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών βασίζονται στην απόκτηση προσόντων για να μπορέσει μετά ο... Πρέπει όμως αυτή η παλιδρόμοι, αυτές οι ρίζες καλύτερα θέλετε, γιατί ε, η λέξη roots σημαίνει και τα δύο στα αγγλικά τουλάχιστον ακουστικά για το διερμηνέα, ε, έχουν ε, λοιπόν το, την ανάγκη να ξεπεράσουν τα σύνορα. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέες, νέους δρόμους ή νέες ρίζες για να αποκτήσουν προσόντα οι άνθρωποι, να έχουν μια ποιότητα για τη ζωή τους, να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια οικονομική ε, δραστηριότητα. Τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ε, εκπαιδευτικών συστημάτων αρχίζουν να ότι Οι χώρες μέλη αποφασίζουν για την οργάνωση και για το περιεχόμενο των συστημάτων εκπαίδευσης. Όμως η ευρωπαϊκή συνεργασία είχε θετική και ισχυρή ε, επίπτωση, επιρροή στους, στα συστήματα αυτά, έχει ενισχύσει την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση, για, δίνοντας τις ενδείξεις για να προωθήσουν την, τον, ε, την, την κοινωνική συμπερίληψη. Το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χώρες μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι ζήτησαν από το ΣΕΤΕΦΟΠ να εκτελέσει τα καθήκοντα αυτά. Εγώ ο ίδιος προσωπικά ως διευθυντής του ΣΕΤΕΦΟΠ έχω εμπειρία για το πώς η γνώση που αναπτύσσει ο ίδιος της ΕΤΕΦΟΠ και την μοιράζεται με τις χώρες μέλη μπορούν να, ε, μπορεί να βοηθήσει να συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων προσόντων μέσα από τα εκπαιδευτικά συστήματα. Πρέπει να βοηθήσουμε να εξασφαλιστούν οι προσπάθειες στο ευρωπαϊκό επίπεδο να φτάσουν στους σωστούς πολλαπλασιαστές στο εθνικό επίπεδο, να δημιουργηθούν δηλαδή σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα ανταποκρινόμενοι και στους στόχους που είχε θεσπίσει ο Σεντεφόπ το 2004 και φέτος. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους και τις χώρες μέλη, εργάζεται ο Σεντεφόπ για να αναπτύξει την γνώση για τους νέους και για τους ενήλικους. Το 2014 δώσαμε υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Εκπαιδευτική Κατάρτιση, που είχε μεγάλη σημασία συνήλθαν οι χώρες μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι σε ένα φόρουμ για την ε, μαθητεία, δηλαδή για να δοθούν ε, θέσεις μαθητευομένων στους νέους. Το 2015 θα συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή και για άλλες χώρες, Σλοβενία, Ελλάδα και Ιταλία. Εργαζόμαστε επίσης για να αναπτύξουμε ευρωπαϊκά εργαλεία για να παρακολουθεί την εξέλιξη των συστημάτων, ε, γιατί Όλα τα συστήματα εκπαίδευση έχουν σημασία. Η κινητικότητα επίση για την μάθηση έχει πολύ μεγάλη σημασία και βεβαίω όλα αυτά πρέπει να συνοδεύουν το άτομο διαβίου. 36 χώρε αναμένεται μέχρι τα τέλη του 2015 να έχουν συνδεθεί με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προσόντων, επιτρέποντας έτσι και σε χώρες μέλη και στις ε, επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τα σχετικά δίκτυα. Ο ΣΕΝΤΕΦΟΠ θα συνεχίσει να εργάζεται και να υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή. Πέρσι ο ΣΕΝΤΕΦΟΠ εξέδωσε μία από τις πρώτες επιθεωρήσεις για την αξιολόγηση της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης έξω από τον δημόσιο τομέα και θα προχωρήσει στην αξιολόγηση και τον επόμενο χρόνο. Έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο εγγράφων διαθέσιμο σε 27 γλώσσες έτσι ώστε να δείξουμε στον κόσμο τις βάσεις των γνώσεων που συμβάλλουμε στην ανάπτυξή τους. Από τότε που ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή το 2005 έχουν δημιουργηθεί 47 εκατομμύρια ε, βιογραφικά επιγραμμικά. Για να υπάρξει λοιπόν η συνοχή μεταξύ αρχών και εργαλείων χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσπάθεια ήδη για το 2015 και χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό σύστημα credit για την εκπαίδευση, για να φτάσουμε στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα που προτείνει με τις συστάσεις του το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεργαζόμαστε επίσης για την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων και των εθνικών και της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Χρειάζονται προσόντα που να ακολουθούν τις τάσεις της αγοράς και αυτά είναι σημαντικό χαρακτηριστικό όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων. Φέτος ο ΣΕΤΕΦΟΠ θα ενημερώσει την πανευρωπαϊκή εστίαση και ανάλυση για κάθε χώρα μέλος. Θα συνεχίσει να συζητεί τις προκλήσεις που απαιτείται να αντιμετωπιστούν για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας. Έχουμε εξετάσει και το έγγραφο του παγκόσμιο Φόρουμ που λέει ότι πρέπει και παρουσιάστηκε στον Ταβό πέρσι ε, για να προσαρμοστούν τα προσόντα στις ανάγκες των αγορών. Η συζήτηση και η συμφωνία για ένα κοινό όραμα για το τι θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα θα βοηθήσει στην επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε μια δύσκολη περίοδο που θα ακολουθήσει την οικονομική κρίση. Βέβαια, οι πόροι είναι περιορισμένοι και ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος λόγω της ανεργίας και λόγω του ότι και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν ακολουθούν πάντα τις πραγματικότητες των αγορών εργασίας. Ο Σεντεφόπ θα συνεχίσει να συμβάλλει στην συζήτηση αυτή και φέτος με την έκθεση που θα εκδώσει ισχυρότερη επαγγελματική κατάρτιση για καλύτερη ζωή που θα εξετάσει την πρόοδο της μεταρρύθμισης των εκπαιδευτικών συστημάτων στις χώρες μέλη. Όμως, για να φτιάξουμε σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα σημαίνει επίσης ότι για να ωφεληθούν οι πολίτες από τα συστήματα αυτά και αυτό σημαίνει βέβαια ακόμα περισσότερα αιτήματα απέναντι στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Ο ΣΕΝΤΕΦΟΠ πρέπει λοιπόν να συμπεριλάβει κάποιες πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν ξεχωριστά, όχι μόνο ευρωπαϊκά εργαλεία, αλλά και γενικότερα που πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των αγορών, ξαναλέω. Αναλαμβάνει ο ΣΕΤΕΦΟΠ νέα καθήκοντα, προσφέρει περισσότερες πληροφορίες και αναλύσεις εξειδικευμένες για κάθε χώρα μέλος και υποστηρίζει συγκεκριμένα χώρες ή και ομάδες χωρών. Ολοκληρώνοντας, ο ΣΕΤΕΦΟΠ επιζητεί την συνεχιζόμενη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έργο του. Ο ΣΕΝΤΕΦΟΠ βεβαίω είναι διατεθειμένος να προσφέρει η αδίποτε πληροφορία είναι απαραίτητη για να υποστηριχθούν οι συζητήσεις και οι γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο συγχρονισμός της αξιολόγησης των συστημάτων θα σημαίνει πάντα πρόοδο. Όμως η ίδια η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία διαβίου. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των πολιτών της Ευρώπης μέσα σε ένα διαφοροποιημένο περιβάλλον. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες από τις οποίες θα ωφεληθούν οι ίδιοι οι πολίτες και για την προσωπική τους και για την οικονομική τους ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγο στον κύριο Μενέντε Βαλντέ, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωση και Εργασία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. όπως μας είπε ο Διευθυντής Καλέγια, ε, είναι 40 ετών το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και εμείς Έχουμε λίγους μήνες διαφορά με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και εμείς θα γιορτάσουμε τα 40 χρόνια φέτος. Είναι 40 χρόνια λοιπόν τα χρόνια ζωής των ευρωπαϊκών οργανισμών. Μερικοί βέβαια είναι νεότεροι, γιορτάζουν μόνο μια εικοσαετία, αλλά Θα θέλαμε να παρουσιάσουμε το έργο των οργανισμών μας στην Επιτροπή με λίγες λεπτομέρειες, γιατί το έχουμε ξανακάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Ε, για τις δραστηριότητές μας για το 2014 υπάρχει το λεπτομερές έγγραφο. Υπάρχει επισκόπηση για το 2015 με τους δείκτες των επιδόσεών μας, τα έχετε λάβει με email και υπάρχουν και όλα τα link, ε, οι σύνδεσμοι για τα έγγραφα που ε, χρησιμοποιούνται ως τεκμηρίωση. Δεν θα ήθελα λοιπόν εδώ να είμαι διεξοδικό στην παρουσίαση, απλώς να πω ότι το 2014 η Eurofound παρουσίασε 1.225 δημοσιεύσεις, εφαρμόσαμε 90, εκτελέσαμε 99,7% του προπολογισμού μας, με όσα μας ενέκρινε η Δημοσιονομική Αρχή, Κοινοβούλιο και ε, Συμβούλιο και αξιοποιήσαμε το προσωπικό μας κατά 99%. Ε, προηγουμένως, η γνώση μας έχει χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον 328 έγγραφα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέρος της αποστολής μας για την παροχή πληροφοριών προκειμένου να βελτιώσουμε και να σχεδιάσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας για τους τομείς του τους κοινωνικούς και τις διαβίωσης. 43% ε, ε, περισσότερα φέτος και το 36% είναι έγγραφα που αφορούν το Κοινοβούλιο. Έχουμε εξακολουθήσει το έργο μας σε τέσσερις ε, πολιτικές προτεραιότητες που συμφωνήθηκαν βάσει του τετραετούς προγράμματος και θα τις αναφέρω πολύ σύντομα. Να δείτε Ποιε είναι από τις βασικές μας δράσεις σε αυτόν τον τομέα. Ξεκινώντας με τον τομέα της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργία. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα του Eurofound. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε προς αυτό το σκοπό, στους τομείς της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, των μικρομεσαίων ή στις επιπτώσεις του χάσματος απασχόλησης των δύο φύλων, τη χαμηλή δηλαδή συμμετοχή στην αγορά εργασίας των γυναικών. Αυτό ξεκίνησε ήδη νωρίτερα, θα συνεχιστεί και φέτος η μελέτη του θέματος για να πετύχουμε τους στόχους της ίσης εκπροσώπηση των φύλων στην αγορά εργασίας βάσει της στρατηγικής του 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε και τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας όπου έχουν πετύχει για να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία τους από τα κράτη-μέλη που έχουν ε, ε, προβλέψει το κόστος, ε, τον περιορισμό του κόστους για, το, για τη μισθολογική εξίσωση και κοιτάζουμε πώς τα κράτη-μέλη μπορούν να τα εφαρμόσουν αυτά κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, παρομοίως, ε, το ίδιο κάνουμε για την νεολαία. Ε, κοιτάζουμε την αποτίμηση πολιτικών όπως την ε, στήριξη των εταιριών για νέους επιχειρηματίες αλλά εξερευνώντας και άλλους τομείς που αφορούν την νεολαία, με την ανεργία των νέων και την απασχόληση των νέων, την κοινωνική τους ένταξη και με ιδιαίτερη μέρημνα στην υλοποίηση της εγγύησης ε, του μηχανισμού για την εγγύηση των νέων ή την ε, ε, ένταξη των νέων. Ο δεύτερος τομέας ενδιαφέροντος είναι η ποιότητα εργασίας και οι συνθήκες εργασίας. Η αγορά εργασία είναι ένα από, τα βασικά, ένα από τα βασικά θέματα έρευνας του Eurofound της τελευταίας δεκαετίας. Θα ξεκινήσουμε επισκέψεις επιτόπιες και συνεντεύξεις ήδη σε λίγες ημέρες με 4.000 Ευρωπαίους πολίτες όπου θα τους ρωτήσουμε για τις συνθήκες εργασίας τους. Θα κάνουμε μια νέα αξιολόγηση της κατάστασης για την ποιότητα της εργασίας και των ε, θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, αλλά θα διερευνήσουμε και από την άποψη του κόστου ζωής ποιες είναι οι συνθήκες που μπορούν ε, να κάνουν την ε, διαβίωση ελκυστική. Δηλαδή πώς οι θέσεις εργασίας θα προσελκύσουν ανθρώπους και θα τους κάνουν να μείνουν πιο μεγάλο διάστημα σε μια θέση. Ε, τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας αυτών και τι, πώς μπορούν να επηρεάσουμε τις σχετικές πολιτικές. Αυτά θα μας απασχολήσουν. Άλλες δραστηριότητες που θα προσπαθήσουμε να τις, ε, με αυτές να εμπλουτίσουμε διάφορες πολιτικές όπως το ευέλικτο σύστημα ε, για την ευέλικτη απασχόληση στη διάρκεια του κύκλου ζωής, η ενδιάμεση αναθεώρηση για να μπορεί κανείς να αλλάξει πορεία επαγγελματική εφόσον το θέλει και ε, για την κατοχή θέσεων εργασίας που να είναι πιο ε, μακροπρόθεσμες. Τρίτος τομέας ενδιαφέροντος στην καρδιά του μηνύματος του Πρόεδρου Γιούνκερ, δηλαδή ανάκαμψη του κοινωνικού, αναθέρμανση του κοινωνικού διαλόγου. καθοριστικός τομέας ενδιαφέροντος για το Eurofound. Βλέπουμε το μεταβαλλόμενο σύστημα των ε, κοινωνικών και εργασιακών σχέσεων και κοιτάζουμε γιατί ε, δεν υπάρχει ε, συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην οικονομική διακυβέρνηση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αλλά και την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Κοιτάζουμε διαφορετικά στοιχεία και τη διάρθρωση του ευρωπαϊκού με το εθνικό επίπεδο λόγω χάρη στα Συμβούλια Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κοιτάζουμε τα σημεία κλειδιά και τα θέματα κλειδιά για την αλλαγή στις αμοιβέ λόγου χάρη, το μηχανισμό εξίσωσης των αμοιβών ή τη μελέτη του χρόνου εργασίας. Τέλος, η ποιότητα ζωής και οι κοινωνικές πολιτικές. Συνεχίζουμε να μελετούμε ένα πρόγραμμα για την πρόθεση της κοινωνικής κινητικότητας στην Ευρώπη και για τις δημόσιες υπηρεσίες, κάτι που είναι κέρια σημασία για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και την, ε, το κοινωνικό μοντέλο. Ε, είναι σημαντικό για τη σχέση εμπιστοσύνη των πολιτών προ τα θεσμικά του όργανα. Αυτό αυτή τη στιγμή, όπω βλέπουμε, ε, δοκιμάζεται στου δύσκολου καιρού που έχουμε γνωρίσει από την αρχή τη κρίση το 2008. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε τα διαφορετικά έγγραφα, απλώς μια σύντομη μνήα σε κάποια στοιχεία που εδώ συζητάτε, την δημιουργία της πλατφόρμας για τις συνθήκες εργασίας. Αυτός είναι ένας τομέας όπου έχουμε αναζητήσει τρόπους να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα της εργασίας και να δημιουργήσουμε μια τράπεζα δεδομένων για γνώσεις. Αυτό είναι ένα από τα βασικά μελήματα του Eurofund και να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το μέλλον της μεταποιητικής βιομηχανίας. Εδώ μας ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Grow και ελπίζουμε να υπογραφεί συμφωνία σχετικά σύντομα θα προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας ως προς τις επιπτώσεις στην απασχόληση των βιομηχανικών πολιτικών και τη διερεύνηση διαφορετικών υποθέσεων για την επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης ε, με θέματα όπως η η μεταφορά των εταιριών, η μετατόπιση τους ή η επιστροφή τους προς την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, η διάσταση της ισότητας των φύλων και η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό το πρόγραμμα θα κρατήσει τουλάχιστον μια τριετία και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζοντας ότι περισσότερες πληροφορίες θα μας έρθουν από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεχίζουμε την ε, συνεργασία με την Επιτροπή σας, με τις συμβουλές που γνωρίζετε, με τις γονικές άδειε, το χρόνο εργασία, ε, την απασχόληση στις μικρομεσαίες και θα αρχίσουμε να συζητούμε ήδη αυτό το μήνα την προεργασία του τετραετούς μας προγράμματος για το 2017 2020. Εδώ θα εκτιμούσαμε την ε, συνεισφορά των πολιτικών ηθινόντων και θα επιστρέψουμε για να μας πείτε ποιες είναι οι, ενδια... οι μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές σας. Πού πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμβάλλει ο Γιώργο Φάρα στον σχεδιασμό πολιτικής. είτε στην, στην Επιτροπή Απασχόλησης του Κοινοβουλίου, είτε σε ποιο άλλο φόρουμ θεωρείται κατάλληλο. Ξεκίνησα αναφερόμενο στα 40 χρόνια ζωής μας να αναφερθώ και να πω ότι είναι 40 χρόνια λειτουργία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Εμεί θα είμαστε ο συντηρητικό οργανισμό για του 42 οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Μαρτίου και θα, ασχολούμαστε με τη, θα ασχοληθούμε με τη συζήτηση του μέλλοντο των Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Αυτό ο συντονισμό θα μα απασχολήσει με νέε ενδεχόμενε διαδικασίε διαχείριση. Ε, θα ξανάρθουμε στην Επιτροπή σας για την απαλλαγή και ε, εκτιμούμε ότι οι εξειδικευμένε επιτροπές που γνωρίζουν το έργο μας όπως η δική σας μπορούν να συνεργαστούν αλλά το ίδιο ελπίζουμε και για την Επιτροπή Προπολογισμού και Ελέγχου των Προπολογισμών. Όλες οι εξειδικευμένες επιτροπές μας ενδιαφέρουν από την πλευρά της συνεργασίας, η θεσμική επίσης διάσταση του έργου μας. Γι' αυτό επιδιώκουμε τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Για τα επόμενα βήματα Μια θεσμική ομάδα εργασίας θα συζητήσει το μέλλον των οργανισμών. Το δίκτυο των οργανισμών αντιπροσωπεύει το 20% του προσωπικού των Ευρωπαίων εργαζομένων, μόνο 0,6% του προπολογισμού, αλλά είμαστε καθοριστικής σημασίας για το θεσμικό αρχιτεκτόνημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είμαστε πλήρως υπόλογοι σε αυτό το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Κρίστα Σέντλατσεκ, που είναι Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Εγώ εκπροσωπώ εδώ πέρα έναν από τους πιο νέους οργανισμούς με την Μαντλίν. Του χρόνου κλείνουμε 20 χρόνια. οργανισμός μας, ο OSHA και θα σας παρουσιάσω το έργο μας το 2014, αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε το 2015 και ελπίζουμε να συνεχίσουμε και να γιορτάσουμε κι εμείς, ίσως όχι υπό τη δικιά μου διεύθυνση, αλλά κι εμείς να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια του ΩΣΑ. Άρχισε το 2014 με ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας 2000 με 2020 με έξι τομείς στρατηγικής σημασίας. Έχουμε ήδη αρκετή εμπειρία. Προσπαθούμε να προκαταλάβουμε τις αλλαγές, να δουλέψουμε πάνω σε αυτές, να βρούμε εργαλεία που βοηθούν τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις στην διαχείρισή τους. Άλλο στόχος μας είναι η συνειδητοποίηση του κόσμου, η δικτύωση. Χρησιμοποιούμε δηλαδή πόρους από ολόκληρη την Ευρώπη προκειμένου να συλλέγουμε πληροφορίες στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Έχουμε και την δικτύωση και την επικοινωνία. Θα αρχίσω λοιπόν με μια εμβληματική μας προσπάθεια που είναι να έχουμε υγιεινούς χώρους εργασίας. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια εκστρατεία προκειμένου να καταπολεμήσουμε το στρες στους χώρους εργασίας. Για δύο χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα αυτό του άγχου στους χώρους εργασίας και τους κινδύνους τους ψυχολογικούς και κοινωνικούς. Μια από τις κύριες δραστηριότητες μας είναι η συνειδητοποίηση του κόσμου και η ενημέρωση στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους, στους κοινωνικούς εταίρους και σε άλλους σημαντικούς παράγοντες. Έχουμε ένα τριμερές συμβούλιο το οποίο αποφάσισε το θέμα αυτό του άγχους και τους κινδύνους τους κοινωνικούς και τους ψυχολογικούς να το κάνει εκστρατεία ακριβώς γιατί διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο ότι 50 με 60% από τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους αυτό οφείλεται στο άγχος που έχουν στην εργασία. Το ίδιο ισχύει και για την πρόορη σύνταξη. Κάτι που καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο κόστος για την κοινωνία. Είναι κάπου 3% του ΕΠ. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Έχουμε αναπτύξει υλικό για την εκστρατεία μας, ιστότοπους και άλλα υλικά σε 24 γλώσσες και ό,τι μήνυμα και αν στέλνουμε είναι σαφές ότι οι κίνδυνοι αυτοί οι κοινωνικοί και ψυχολογικοί μπορούν να εκτιμηθούν, να υπολογιστούν και να αντιμετωπιστούν. Έχουμε αναπτύξει επίσης μια ευρωπαϊκή εκστρατεία που το ονομάζουμε ECAP. Είναι ευρωπαϊκή, ένα πακέτο ευρωπαϊκής εκστρατείας αρρωγής συμπεριλαμβάνουμε διάφορες δραστηριότητε σε εθνικό επίπεδο και στις 28 χώρες μέλη. Και αυτό το κάνουμε σε στενή σχέση με τα εθνικά σημεία επαφής που έχουμε, τα focal points. Έχουμε ήδη οργανώσει 20 εκδηλώσεις εμείς και επιπλέον τον Οκτώβριο οι χώρες μέλη από μόνες τους οργάνωσαν άλλες τόσες εκδηλώσεις. Προσλάβαμε επίσης πάνω από 100 συνεταίρους κατά κάποιο τρόπο στις εκστρατείες αυτές από τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους οι οποίοι θέλησαν να στηρίξουν την εκστρατεία αυτή μέχρι και το 2015 και οργανώνουν και αυτοί εκδηλώσεις και για να σας δώσω κάποια παραδείγματα είναι διάφορες επιχειρήσεις που συμμετέχουν, η Χάνικεν, η Toyota, η Ζήμεν, η Σπιρέλη και πολλές άλλες. Για πρώτη φορά έχουμε και έναν ηλεκτρονικό οδηγό. Είναι μια εύκολη εφαρμογή η οποία προσφέρει πληροφορίες σε όλους. Είναι δωρεάν. Και σε αυτόν τον οδηγό εξηγούμε τι είναι το άγχος, το στρες, ποιες είναι οι συνέπειες, ποιες είναι οι αιτίες και πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί, να αντιμετωπίσει το άγχος. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω για τις επιχειρήσεις. Έχουμε τις διάφορες εκδοχές και στις 28 γλώσσες και συμπεριλαμβάνουμε και την εθνική νομοθεσία και εθνικές πηγές. Μέχρι τα τέλη του 2015 μαζί με τους εταίρους μας θα οργανώσουμε και άλλες εκδηλώσεις. Έχουμε ένα βραβείο της πρακτικής από κοινού με τη Λετωνική Προεδρία, όπου θα βραβεύσουμε τις πιο πετυχημένες επιχειρήσεις, που μπόρεσαν δηλαδή με επιτυχή τρόπο να αντιμετωπίσουν το στρες στους χώρους εργασίας. Και τέλος, θα έχουμε στο Μπιλμπάο στα τέλη της χρονιάς ε, κάποιο είδου διάσκεψη για να κλείσει η εκστρατεία αυτή του 2015 λοιπόν θα ολοκληρωθεί η εκστρατεία αυτή και συζητάμε ήδη με το Διοικητικό μας Συμβούλιο το θέμα της επόμενης εκστρατείας που θα έχουμε για τα έτη 2016 και 2017. Αποφασίστηκε ότι θα έχει να κάνει με τον ε, πιο ηλικιωμένο πληθυσμό στην εργασία, με την γύρανση δηλαδή δουλεύοντας. Μας ενδιαφέρει η υγεία και ασφάλεια όλων των εργαζομένων Ήδη από το 2013 έχουμε μία έρευνα μετά από απόφαση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη δουλειά την ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Όσα να κάνει δηλαδή αυτή την έρευνα. Στα πλαίσια αυτά και εμείς προσπαθούμε να αναλύσουμε τις δραστηριότητε των χωρών μελών, να αξιολογήσουμε τις προϋποθέσεις για να έχουμε υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας για τα πιο ηλικιωμένα άτομα. Συλλέγουμε εμπειρίες και θα παρουσιάσουμε και τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς επίσης και προτάσεις για να βοηθήσουμε τους πολιτικούς που αποφασίζουν τελικά για τις αντίστοιχες πολιτικές. Ήδη σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών μελών για το πώς αντιμετωπίζουν την ασφάλεια και την υγιεινή, για τον όλο και περισσότερο γυράσκοντα ε, εργαζόμενο πληθυσμό. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν διαφορές σε όλες τις χώρες μέλη. Στα μέσα του 2015 θα οργανώσουμε μια διάσκεψη και ελπίζω να έχουμε και εσάς μαζί μας για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής η οποία θα δημοσιευθεί στα τέλη του 2015 θα αποτελέσει τη βάση για τις συστάσεις που θα κάνουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το συστήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έρχομαι τώρα στα μέσα που έχουμε για την διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Ξέρετε ότι έχουμε μία έρευνα online για την ε, αξιολόγηση κινδύνου, το OIRA. Είναι δωρεάν Στηρίζει την αξιολόγηση λοιπόν των κινδύνων στους χώρους εργασίας όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια. Συμμετέχουν 14 χώρες τώρα που έχουν αναπτύξει παρετέρω τόιρα, δηλαδή στις γλώσσες τους έχουν συμπεριλάβει την εθνική τους νομοθεσία, αλλά βέβαια και τις Επιτροπές Κοινωνικού Διαλόγου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ήδη αρχίσει να δημοσιεύουμε και μία στρατηγική ενόψη του 2006 για να κοινοτοποιηθούν περισσότερες χώρες και περισσότεροι κλάδοι να συμμετάσχουν στο εργαλείο αυτό το online, το OIRA. Από ό,τι φαίνεται είναι μια πραγματική επιτυχία. Τα δύο τελευταία χρόνια δηλαδή τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα επιτυχή. Και έτσι έρχομαι και στο Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας, σχετικά με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση πριν από λίγο καιρό. Αναφέρεται συχνά εκεί και ο οργανισμός μας. Και τώρα το 2015 και μέχρι το 2020 θα έχουμε ρόλο κλειδί στην εφαρμογή αυτού του πλαισίου πολιτικής, όχι μόνο βάσει του όιρα, αλλά και βάση της έρευνάς μας, την οποία θα αναφερθώ αργότερα. Άλλες δραστηριότητες που θα κάνουμε το 2015, αλλά και 2016 και 2017, είναι ότι αρχίσαμε ήδη ένα μεγάλο σχέδιο για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε πολιτικές, βέλτιστες πρακτικές και έρευνα για το υπόβαθρο αυτού του θέματος μέσα στους επόμενους μήνες. Έτσι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε παρετέρω για τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε αρχίσει προγράμματα για το βάρος από τραυματισμούς ε, και ασθένειες. Εξετάζουμε και το θέμα των επενδύσεων που δεν είναι αρκετές συχνά για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας. Ελπίζω σε μερικούς μήνες να μπορέσουμε να σας υποβάλουμε και δεδομένα από την δεύτερη έρευνά μας, ευρωπαϊκή έρευνα, για τους αναδυόμενους νέους κινδύνους της επιχειρήσης. Επικεντρωνόμαστε τώρα ήδη σε επιχειρήσεις που δουλεύουν με πέντε ή περισσότερους εργαζόμενους. Στο μέλλον όμως θα συμπεριλάβουμε και πιο μικρές επιχειρήσεις. 36 ε, χώρες, καλύπτουμε όλους τους κλάδους και δουλεύουμε και βάσει μιας καλύτερης μεθοδολογίας. Θα μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε στοιχεία τα οποία να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να υιοθετούν προληπτικά μέτρα. Θα αναφέρουμε επίσης τις ανάγκες των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους, με τον κλάδο στον οποίο απασχολούνται, την τοποθεσία τους και επικεντρωνόμαστε επίσης σε ειδικό εργατικό δυναμικό που είναι πιο ηλικιωμένοι. Πολύ σύντομα Ελπίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης να μπορέσουμε να σας τα παρουσιάσουμε αυτά για να έχουμε και τη δικιά σας τη άποψη. Στο Wikipedia τώρα και στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας και εκεί έχουμε αρχίσει κάτι. Έχουμε εκεί ενημέρωση, που την ενημερώνουμε μάλιστα κάθε τόσο, και θα αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία ενημέρωσης όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και πέρα από την Ευρώπη. Συμμετέχουμε επίσης στις δραστηριότητε ΕΠΕ και στο πρόγραμμα γυτνίασης που θα αρχίσει σύντομα. Τέλος, κάναμε μια έρευνα με 3.000 που απάντησαν προκειμένου να μας πούν την άποψή τους για τη δουλειά μας. Οι απαντήσεις είναι πολύ θετικές. Νομίζω ότι είναι ικανοποιημένοι. Κυρίως το μήνυμά τους είναι ότι από εμά παίρνουν πληροφορίες που δεν μπορούν να βρουν σε άλλες πηγές. Καλύπτουμε δηλαδή ένα κενό και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που είναι πολύ θετικό για μας. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι πολύ χρήσιμες για μας, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον, πώς θα κινηθούμε και πώς θα συνεργαστούμε με τους, με τους κοινωνικούς εταίρους, μαζί σας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τώρα μένει να λάβει το λόγο η κυρία Σέρμπαν, που είναι διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Εκπαίδευσης, ETF. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πάντοτε αποτελεί τιμή να εμφανίζομαι ενώπιόν σας και βεβαίως να προσπαθήσω σε λίγα λεπτά να εξηγήσω ποια θεωρώ ότι είναι τα ισχυρά σημεία του οργανισμού μας και βεβαίως να λάβω από εσά τις κατευθύνσεις για το τι να συνεχίσουμε να κάνουμε. Όπως λέχθηκε και δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα ατζέντα. Ε, ορισμένοι μιλούν ούτε, ούτε, ούτε ηλικία, γιατί εδώ έχουμε οργανισμού που έχουν ήδη μια ηλικία 40 ετών, εμεί έχουμε μικρότερη. Η συνεργασία των οργανισμών μα μπορεί να προσφέρει καλύτερη υποστήριξη στο δικό σα έργο και όπω είπαν και οι προηγούμενοι συναδελφοί μου και εμεί είμαστε διατηθειμένοι να είμαστε στη διάθεσή σα δηλαδή για, ε, με τον οργανισμό μα για να σα υποστηρίξουμε. Είπα τον Νοέμβριο του 2014 ότι το ETF δημιουργήθηκε μια χρονιά που γιορτάζαμε 25 χρόνια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και ήταν μάλιστα και η χρονιά της εκατονταετίας του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου, 2014 δηλαδή. Εμείς δουλεύουμε για τον άνθρωπο, για να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα μπορεί να συνεργαστεί με τις γειτονικές της χώρες σε ισότιμη και ισοδίκαιη βάση. Σήμερα ενώπιόν σας προσπαθώ να εξηγήσω ότι και το 2015 η εντολή μας θα παραμείνει ίδια. Θα ήθελα να σας εξηγήσω με μία από τις δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker που αναφέρεται σε ισχυρότερη παγκόσμια δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως αποφασίσατε εσείς αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει ο τέταρτος τίτλος, Heading 4, Global Europe στον κοινοτικό προϋπολογισμό και εμείς κάνουμε κάθε τι που περνάει από το χέρι μας για να συμβάλλουμε στον προσανατολισμό της συνεργασίας προς τις χώρες που καλύπτει η εντολή μας. Αυτά που περιλαμβάνει η σχετική προτεραιότητα είναι ότι υπάρχει ανάγκη συστηματικής προβολής προς τα, προς τα έξω των εσωτερικών πολιτικών για να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί στόχοι πολιτικής είναι παρόντες, ορατοί και επηρεάζουν την παγκόσμια σκηνή. Για να το κάνουμε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει σημαντικότερος ε, παίκτη στο παγκόσμιο επίπεδο θα συνεχίσει να εφαρμόζει δημοκρατικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, να διατηρεί το κράτος δικαίου, να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, να αναπτύσσει θεσμικές ικανότητες και μια λειτουργική ε, δημόσια διοίκηση στις χώρες αυτές που είναι στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Τουρκία, χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και Νότιας Γειτονίας και χώρες που συμμετέχουν μαζί μας στην προσπάθεια αναπτυξιακής βοήθειας. Το 2015 είναι το, έτος, το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό να λεχθεί σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση στον τομέα της δικής μας δουλειάς είναι να πούμε ότι ο κόσμος ολόκληρος αντιμετωπίζει μια διαρθρωτικά μεγάλη ανεργία και υποαπασχόληση. Βαθιά πολιτική και κοινωνική αστάθεια που προκαλεί καμιά φορά απρόβλεπτες και πολύ δύσκολο να τις διαχειριστεί κανείς μεταναστευτικές κινήσεις και προσθέτει σημαντικό αριθμό προσφύγων που κινούνται όχι αποκλειστικά μεταξύ των χωρών εταίρων μας αλλά και προς την Ευρώπη. Υπάρχει και μια βαθιά εισοδηματική ανισότητα την οποία επίσης παρατηρούμε παγκόσμια. Δυστυχώς η οικονομική κρίση μας έβαλε σε μια θέση που βλέπουμε να συμπιέζεται η μεσαία τάξη των αναπτυσσόμενων χωρών. Όταν μιλούμε όμως για αυτό το παγκόσμιο στοιχείο που είναι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, Διαπιστώνουμε επίσης ότι και στις χώρες εταίρους μας η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει σε μια πόλωση των εισοδημάτων. Και αυτό παρατηρούμε τώρα, γι' αυτό παρατηρούμε τώρα, πολύ βαθιά φτώχεια που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές. Όμως το εμπόριο, το περιβάλλον και η ανάπτυξη είναι παγκόσμιες διαστάσεις εξορισμού. Όμως στην Ευρώπη έχουμε αρχίσει ήδη κάποιες πρωτοβουλίες που μπορούν να προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις μας να γίνουν διεθνείς. Μικρές και μεσές επιχειρήσεις για παράδειγμα. Και η πρόθεση που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι για να δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να δημιουργήσουν απασχόληση, να μπορέσουν να προβούν σε συναλλαγές δηλαδή και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πρωτοβουλία επίσης η οποία θα επιστρέψει σε εσά και μιλώ εδώ για την γαλάζια κάρτα που θέλω να σας αναφέρω και λίγο αργότερα. Η Ευρώπη όμως για να γίνει παγκόσμιος παίκτη δεν επιτρέπεται να λησμονήσει ότι έχει το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού. Για την ώρα έχει μόλις το 10% της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, αλλά έχει και καλά νέα, διότι η Ευρώπη δαπανά το 50% των κοινωνικών δαπανών. Δηλαδή το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο θα συνεχίσει να επηρεάζει τον υπόλοιπο κόσμο. Διότι εάν η Ευρώπη συνεχίσει έτσι αποτελεί το όραμα για όλες τις χώρες εταίρους και η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι μοντέλο για την ε, περαιτέρω εξέλιξη στο κοινωνικό τομέα. Λέχθηκε επίσης πρόσφατα από τις επιτρόπους που ήλθαν εδώ για να τους ακούσετε στις ακροάσεις τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Ευρώπη είναι και ο μεγαλύτερος δωρητής με την έννοια ότι προσφέρει το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης και υποστήριξης στις χώρες του κόσμου. Είναι λοιπόν ο μεγαλύτερος δωρητής και η Ευρώπη θα ήθελε να μην είναι πλέον αυτός που πληρώνει, ο payer δηλαδή, αλλά να γίνει player, να είναι πραγματικός παίκτη στην παγκόσμια σκηνή. Εσείς αποφασίσατε να παίξει το ρόλο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτή η ήπια δύναμη στις εξωτερικές σχέσεις αλλά βέβαια το ανθρώπινο κεφάλαιο μόνο του δεν μπορεί να τα καταφέρει. Χρειάζεται και το κοινωνικό κεφάλαιο και εκεί ερχόμαστε εμείς και πρόκειται για τον κόσμο, για ανθρώπους. Θα ήθελα τώρα να σας προσφέρω, αν μου επιτρέπετε, μια ξενάγηση στο έγγραφο αυτό για το τι κάνουμε δηλαδή. Πρώτα, ποιο είναι το πιστεύω του ETF και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το μέλλον των πολιτών θα πρέπει να είναι στις ίδιες τους τις χώρες. Γι' αυτό δουλεύουμε με όλες τις χώρες εταίρους μας για να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ανταγωνιστικότητάς τους στις ίδιες τους τις χώρες. Όμως οι ευρωπαϊκές αξίες, ελεύθερη διακίνηση δηλαδή, εφαρμόζονται και στις χώρες εταίρους μας. Αν λοιπόν αυτές οι χώρες θέλουν να προχωρήσουν σε νόμιμη μετανάστευση, μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Όμως το να δουλέψουμε έτσι ώστε να έχουν μέλλον στις ίδιες τους χώρες, αυτό μετριάζει τον κίνδυνο της αυξημένης μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να ενισχύσουμε δηλαδή την ευρωπαϊκή εμπλοκή παγκόσμια. Αυτό που κάνουμε είναι ότι εργαζόμαστε πάνω σε πολιτικές για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου που να εμπνέονται από την εξωτερική διάσταση των εσωτερικών ευρωπαϊκών πολιτικών με πολιτικές για ανάπτυξη προσόντων, ικανοτήτων και συνδυάζουμε την πρόβλεψη για το 2020 με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες του οικονομικού τομέα για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει δουλειά εκεί όπου χρειάζεται και ότι θα υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη που θα οδηγήσει στη δημιουργία απασχόλησης και όχι μονάχα κερδών για τον οικονομικό τομέα. Τα κάνουμε λοιπόν αυτά και εικονογραφώ αυτά που κάνουμε με την περίπτωση της Αλβανίας, χώρα στην οποία όπως και στις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και στην Τουρκία έχουμε κάνει μια προσπάθεια να συνεργαστούμε με τον δημόσιο τομέα για να ενισχύσουμε την ικανότητά του να αντιμετωπίσει τις απαραίτητες πολιτικές και με τα μεσοπρόθεσμα σχέδια δαπανών της χώρας, βάζοντας και ένα σύστημα monitoring, παρακολούθηση δηλαδή για τις πολιτικές αυτές, όπου να λαμβάνει υπόψη και τα αποτελέσματα που μπορεί να επιτύχει. Πρόσφατα, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας είπε σε διεθνή σύσκεψη ότι με τη δική μας συμμετοχή αλλά με δική του απόφαση ήταν σε θέση να αναδιαρθρώσει την κυβέρνησή του, να αναδιαρθρώσει τις δαπάνες του προϋπολογισμού του για ανθρώπινο κεφάλαιο, τις οποίες τριπλασίασε στη βάση ενός οδικού χάρτη, ακολουθεί βεβαίως και όλους τους δείκτες monitoring στην χώρα του και τα Υπουργεία του το αναφέρουν για τους δείκτες monitoring που έχουμε ε, θεσπίσει σε συνεργασία μαζί τους. Εμείς είμαστε πολύ υπερήφανες που καταφέραμε με την σε βάθος γνώση της χώρας μας τι ακριβώς χρειάζεται η χώρα αυτή, η Αλβανία δηλαδή πάντα. Βεβαίως αυτό ήθελε ο Πρωθυπουργό να μπορεί να ανακοινώσει σε ολόκληρη την κοινότητα ότι η Ευρώπη, στη διεθνή κοινότητα δηλαδή, ότι η Ευρώπη του προσφέρει μεγάλη βοήθεια. Βέβαια οι πολιτικές από μόνες τους δεν μπορούν να τα προσφέρουν όλα. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι απαραίτητο κλειδί. Γι' αυτό πιστεύουμε σε μια διακυβέρνηση που να την συνυποστηρίζουν όλοι οι φορείς να είναι συμμετοχικοί, αποτελεσματικοί και να προβλέπει ποιες θα πρέπει να είναι οι σωστές πολιτικές. Και βεβαίως να περιλαμβάνει και το στοιχείο του επιχειρήν, να μην αναμένει από τους άλλους να πούν τι θα πρέπει να γίνει. Σε αυτή τη διακυβέρνηση εμείς συνεργαζόμαστε και με τις κυβερνήσεις και με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους διάφορους τομείς, αλλά και με τις περιφέρειες. Εάν δεν είναι ικανοί οι φορείς αυτοί να παίξουν ένα ρόλο, δεν θα παραμείνουν εταίροι μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό και παρουσιάζουμε σήμερα την εργασία μας εδώ και στην περίπτωση της Ουκρανίας, όπως σας είπα και τον Νοέμβρη, όταν στο Μαϊντάν οι άνθρωποι ζητούσαν την ελευθερία τους, εμείς εκεί συνεργαστήκαμε με όλες τις περιφέρειες της Ουκρανίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο κόσμος αγωνιά για το μέλλον του και εκεί η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει και οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν μαζί μας και εμείς είμαστε διατεθειμένοι βεβαίως να συνεργαστούμε. Το ίδιο για την Τινησία όπου η Αραβική Άνοιξη πρόσφερε πολλά, πολλές προσδοκίες στους πολίτες. Δυστυχώς όμως οι επενδύσεις είναι απαραίτητες, είναι το κλειδί για την παραπέρω πορεία. Όμως δεν, γίνονται, δεν είναι σωστά κατανεμημένες οι επενδύσεις εκεί, διότι σχετικά, συνήθως όλες οι επενδύσεις κατευθύνονται στην πρωτεύουσα. Εκεί συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση της Τινησίας για να προσφέρουμε ίσες δυνατότητες σε όλους τους Τινήσιους πολίτες όπου και να βρίσκονται και να υπάρχει μια συνοχή, μια εδαφική συνοχή που όπως είπα να επιτρέψει σε όλους τους Τινήσιους να έχουν μέλλον είτε στην πόλη τους είτε στην περιφέρειά τους. Και τα κάνουμε αυτά σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα και με τους ανώνυμους αστέρες όλων αυτών των χωρών που μπόρεσαν να μας εξηγήσουν με ποιο τρόπο μπορούν να συνδιαμορφώσουν τις εθνικές πολιτικές, πώς μπορούν να επανέλθουν και να εφαρμόσουν τις εθνικές αυτές πολιτικές. Έχουμε και ορισμένα παραδείγματα στο έγγραφό μας. Μίλησα για το επιχειρήν η μάθηση για το επιχειρήν είναι ουσιώδης για όσα κάνουμε. Μίλησα και για το επιχειρήν μέσα στα οικοσυστήματα όταν μίλησα για την πολιτική, όταν μίλησα για τις κυβερνήσεις που δημιουργούν θεσμούς για το επιχειρήν και εκεί παίζουμε ένα ρόλο και εμείς. Αλλά όλοι μαζί εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε για να δώσουμε την ικανότητα στους ανθρώπους να ασκήσουν περισσότερο την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν θέλουμε όλοι οι πολίτες να γίνουν επιχειρηματίες. Αυτό που θέλουμε να γνωρίζουμε είναι ότι δημιουργούμε μια ανθεκτικότητα και οι άνθρωποι είναι πια ικανοί να προσαρμόζονται στις αλλαγές που σημειώνονται στις πατρίδες τους. Και όπως ξέρετε, για να σας εξηγήσω μια πολιτική που είναι, που είναι εφαρμόζεται και εδώ στην Ευρώπη, είναι το νομοθέτημα για τις μικρές επιχειρήσεις, Small Business Act, και που αυτό το μεταφέρουμε ως αρχή και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και στην Τουρκία και ευχαριστώ να επανέλθουμε να σας εξηγήσουμε ποιε είναι οι βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν από την τελευταία χρήση. Εμείς δουλεύουμε για να προσφέρουμε δυνατότητες στους ανθρώπους είτε να μείνουν στα σπίτια τους αλλά και στην περίπτωση που θέλουν να μετακινηθούν στην Αλοδαπή εφόσον τους επιτρέπεται αν θέλουν να έλθουν στην Ευρώπη θα πρέπει το μήνυμα και ευχαρίστως να σας το εξηγήσω εδώ εδώ στον οίκο της Δημοκρατίας της Ευρώπης ότι χρειάζεται διαχείριση της μετανάστευσης όχι μόνο στη χώρα προέλευσης αλλά και στη χώρα προορισμού και εξακολουθούμε να παρακολουθούμε ότι δυστυχώς οι προσοντούχοι νόμιμοι βέβαια μετανάστες δεν επιλέγουν την Ευρώπη ως πρώτο προορισμό τους και το τίμα που πληρώνει η Ευρώπη θεωρούμε ότι μπορεί να βελτιωθεί για να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία υποφελή κατάσταση μέσω της γαλάζιας κάρτας. Όταν οι πολίτες αυτοί αποφασίζουν να μεταναστεύσουν θα πρέπει να τους δοθεί το δικαίωμα αυτό. Μιλώ πάντα για νόμιμους μετανάστες. Να μεγιστοποιηθεί η διάσταση των προσόντων της μετανάστευσης. Μιλούμε για αυτή τη μετανάστευση γιατί και οι χώρες προέλευσης των μεταναστών δεν κάνουν αρκετά για να τους προετοιμάσουν και κάνουν και πολύ λίγα για να τους πείσουν αυτούς που έχουν μεταναστεύσει για ένα διάστημα να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους και βεβαίω να αναγνωρίσουν τα προσόντα που έχουν αποκτήσει στην περίπτωση, στην αυτή. Για το 2015 είναι το έτος της ανάπτυξης. Είναι βέβαια και το έτος όπου στη διάρκεια της Λετωνικής Προεδρίας και πάλι η ε, σχέση ανατολικής γειτονίας θα τεθεί υπό συζήτηση. και πολύ ευχαρίστως να συζητήσουμε εμείς βάζοντας μέσα και το, κεφα... ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και για να γίνουν οι πολιτικές πιο αξιόπιστες και να λειτουργήσουν υπέρ των ανθρώπων. Θα συνεργαστούμε με τη Λετωνική Προεδρία και στις 3 και 4 Ιουνίου θα ε, διεξαχθεί διάσκεψη με όλες αυτές τις χώρες για τον χειρισμό των θεμάτων αυτών, για το πώς μπορούν να μάθουν από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και θα θέλαμε πολύ να έχουμε και εσά μεταξύ των συζητούντων. Ελπίζω λοιπόν πραγματικά ότι με τα όσα έχουμε αναπτύξει στο έγγραφό μας θα μπορέσετε να προσφέρετε την εμπιστοσύνη σας διότι η απόδοσή μας μιλεί από μόνη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε εμείς. Θα δώσω το λόγο στη Γιούτα Στάινρουκ, συντονίστρια από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ή... Όχι, όχι, να ξεκινήσουμε με εσάς. Ίσως να ξεκινήσουμε με την συνάδελφα του ΕΛΚ. Όχι, θα ξεκινήσουμε με τη Γιούτα. Αντιδράσεις, ερωτήσεις. Παρακαλώ. Στάινρικ, πάρα πολλές ερωτήσεις. Έχω. Αναρρύθμιτες. Δεν θα μπορέσω να τις θες όλες. Αλλά κατά τα Ιωθώτα των τελευταίων ετών θα τις θέσω διμερώς. Πρώτα όμως θέλω να ευχαριστήσω όλους τους οργανισμούς, όλες τις συνεργάτηδες και τους συνεργάτες των οργανισμών. Είμαι έξι χρόνια τώρα ευρωβουλευτής εδώ, στην Επιτροπή Απασχόλησης και όπως το αισθάνομαι εγώ, το αισθάνονται και οι άλλες συναδέλφισες των και συνάδελφοι των σοσιαλδημοκρατών. Χρειαζόμαστε γνώση, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα εργαλεία, να μπορούμε να βασιστούμε στις δραστηριότητες των οργανισμών σας, που είσαστε σημαντικά εργαλεία για τη δουλειά όλων μας. Και είμαι πολύ χαρούμενη που λειτουργεί καλά και η διαδικτύωση μεταξύ σας, μεταξύ των οργανισμών. Και ακούγοντας από τις παρεμβάσεις σας, διαπιστώνω ότι περιλαμβάνεται και το εθνικό επίπεδο και πολύ εντονότερα μάλιστα. Έχω βέβαια πολλά σχόλια για κάθε έναν από τους οργανισμούς. Θα προσπαθήσω βέβαια να συντομεύσω. Πρώτα για τον ΣΕΔΕΦΟΠ. Είστε σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων για την δημιουργία δομών μέσα στην ίδια την Ευρώπη, αλλά και για τη μελλοντική δουλειά. Τι χρειάζεται, δηλαδή τι είδους προσόντα χρειάζονται για το μέλλον. το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την διπλή επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρώπη. Υπάρχει, αλλά δεν αρκεί να αντιγραφεί ένα προς ένα το τι γίνεται ήδη σε ορισμένες χώρες μέλη. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτείνεται λοιπόν. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η πορεία είναι πολύ αργή στις χώρες μέλη υιοθέτηση δηλαδή και εφαρμογή τέτοιων μοντέλων, παρόλο που πολλοί θα ήθελαν να εφαρμοστούν. Τι προτείνεται λοιπόν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη στην περίπτωση αυτή, που βλέπετε να εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα εμπόδια. Βλέπουμε σημαντικές δυσκολίες των χωρών μελών να απορροφήσουν κονδύλια για την πρωτοβουλία για την νεολαία. Πού βλέπετε ότι υπάρχουν τα σημαντικότερα εμπόδια. Στο ίδιο πλαίσιο έχουμε πολλούς και όχι μόνο νέους ή νέες άνεργους στην Ευρώπη. Έχουμε και πολλούς μακροχρόνια άνεργους για μεγάλες περιόδους της ζωής τους. Κάνετε αναλύσεις και για την μετεκπαίδευση και την παραπέρα κατάρτιση αυτών των ομάδων στόχων. Τώρα, Τώρα για τον κύριο Μέντες Βαλτές του Eurofound. Εσείς περιγράψατε διάφορα tools, εργαλεία δηλαδή, και είναι και πολύ ενδιαφέρον αυτό που προτείνεται για την αξιολόγηση της ποιότητας της εργασίας στην Ευρώπη. Μίλησα, μιλούσα μάλλον προ μικρού χρονικού διαστήματος με συνδικαλιστές ενός συγκεκριμένου τομέα και μου είπαν ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, να γίνουν δηλαδή συγκεκριμένες, στοχευμένες αναλύσεις. Εξάλλου, ο κοινωνικός διάλογος χθες είχαμε συνάντηση με Γερμανούς συνδικαλιστές και είναι πολύ καθαρό και από τις δύο πλευρές, και από τους εργαζόμενους και από τους εργοδότες, ότι ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να λειτουργήσει με επιτυχία μόνο εφόσον και οι δύο εταίροι έχουν κάποια δύναμη, εφόσον μπορούν να συζητήσουν, να μαλώσουν και τελικά να καταλήξουν σε λύσεις, αλλά ισότιμα. Με ποιο τρόπο παρακολουθείτε, συνοδεύετε εσείς τον κοινωνικό αυτό διάλογο. Βλέπετε να γίνονται κάποιες πρόοδοι σύμφωνα με τις βέλτιες πρακτικές που έχουμε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχουμε ισχυρές κοινωνικές διασυνδέσεις, ενώ υπάρχουν άλλες χώρες που θεωρούν τους συνδικαλιστές μαφία. Βλέπετε να γίνουν, υπάρχουν εδώ στην Ευρώπη κάποιες συγκρίσιμε εξελίξεις και ποιο θεωρείτε ότι είναι το επιτυχημένο μοντέλο του κοινωνικού διαλόγου, όχι βέβαια μόνο για ολόκληρο τον κόσμο, αλλά πρώτα πρώτα να κοιτάξουμε στην Ευρώπη, δηλαδή να εξαγάγουμε το μοντέλο αυτό στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Βιομηχανική πολιτική ήταν και ένα από τα θέματα για τα οποία μιλήσατε πώς μπορεί ο κοινωνικός αυτός διαλόγος να οδηγήσει στην εκ νέου εκβιομηχάνηση της Ευρώπης. Και κάτι με ενδιαφέρει επίσης πολύ. Με ενδιαφέρουν πολύ και οι αναλύσεις της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι πιο πετυχημένες μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Έχετε παραδείγματα μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας που δεν απέδωσαν αποτελέσματα ή απέδωσαν αρνητικά αποτελέσματα, γιατί και αυτό μπορεί να αποτελέσει δίδαγμα για μας. Για τον οργανισμό όσα το στρες, η κατάθλιψη στον τόπο εργασίας σημαίνει βαρύτατο κόστος για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και βέβαια για τους θυγόμενου αποτελεί πολύ μεγάλη επιβάρυνση. αντιμετωπίζουμε και την πρόκληση ότι το εργατικό δυναμικό είναι όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Πάλι αυτό σημαίνει σημαντικές προκλήσεις για την αργοδάρα εργασία, αλλά και για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας ιδίω. Τι μπορεί να γίνει εκεί. Εδώ στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο διεξάγεται η συζήτηση για το λεγόμενο REFIT, την βελτίωση νομοθεσίας. Εσείς ως οργανισμός εμπλέκεστε στις συζητήσεις αυτές. Σίγουρα αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι χρειαζόμαστε την τεχνογνωσία σας για το έργο μας. Γιατί η προστασία της ε, υγείας και της ασφάλειας των εργατών είναι σημαντική, σημαντικό θέμα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο refit. Μια συγκεκριμένη ερώτηση τώρα για το όιρα. Είναι καλό εργαλείο, εξυπηρετεί μικρές και μέσες επιχειρήσεις. Γνωρίζω ότι σε πολλές χώρες ε, χρησιμοποιείται, σε πολλές οργανώσεις συμφωνείτε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα εργαλεία και όργανα και να αναπτυχθούν τέτοια για μικρές και μέσες επιχειρήσεις. Λυπούμε πολύ που μακρηγορώ τόσο πολύ, ήταν και πολλοί οργανισμοί, λέει η κυρία Στάιν Ρουκ, για τον οργανισμό ETF. Καλά είπατε ότι δεν πρέπει να στρέφουμε τα βλέμματα μόνο προς τα μέσα, αλλά βέβαια και εξαιτία των προβλημάτων και των εξελίξεων, δεν είναι βέβαια μόνο προβλήματα, είναι και, μπορεί να πει κανεί και, και εξελίξεις, γιατί η μετανάστευση έχει και πολύ θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Εκπαίδευση κατάρτιση σημαίνει και εκδημοκρατισμό. Εφόσον προσφέρουμε λοιπόν εκπαίδευση κατάρτιση στι ίδιε τι χώρες αυτές, στι χώρες εταίρου μας δηλαδή, ενισχύουμε και τη δημοκρατία. Αυτό είναι σημαντικό, γνωρίζω και από τη δουλειά μου στην αντιπροσωπεία σχέσεων με τι βαλκανικές χώρες, ότι συμβάλλεται και μέσα σε αυτό το πλαίσιο στην ανάπτυξη και τέτοιων συστημάτων. Και αυτό θα έχει θετικές συνέπειες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις διαπιστώσεις που κάνετε είναι ότι δεν εμπλέκονται αρκετά οι τοπικοί φορείς και ότι συχνά υπαγορεύουν τα αναγκαία προσόντα, τα ποια θα πρέπει να είναι τα αναγκαία προσόντα, οι κεντρικοί φορείς, οι κεντρικές αρχές. Μου φαίνεται μίλησατε για την Τινησία ως παράδειγμα. Πώς μπορούν όμως να ενισχυθούν εκεί οι ρόλοι των κοινωνικών εταίρων και των συνδικαλιστών επομένως. Την ιδέα με το σύστημα της ε, γαλάζιας κάρτας που αναφέρατε μου φαίνεται, αυτή λοιπόν η ιδέα μου φαίνεται σωστή. Κοιτάξτε είναι τέσσερις οργανισμοί, είμαστε πολύ λίγοι ευρωβουλευτές, σωστό είναι να διεξαχθεί κάποιος διάλογος με τους οργανισμούς. Τελειώνω όμως, τελειώνω τώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να εξαγάγουμε τις καλές πλευρές των πολιτικών μας. Uh, Επόμενη ερώτηση στην κυρία Σεντερόβα. Ευχαριστώ για την ε, παρουσίασή σας. Ευχαριστώ όλους μας τους προσκεκλημένους. Είμαι νέα βουλευτής και για μένα είναι πολύ σημαντικό να ε, καταλάβω το έργο σας και να, να αισθανθώ οικειότητα ε, με τα όσα κάνετε. Για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ να ρωτήσω ότι όλες τις μελέτες που γίνονται για την επαγγελματική κατάρτιση μας είπατε ότι εκπονούνται γρηγορότερα ή αργότερα στις περισσότερες χώρες. Όμως πρέπει να εκπονούνται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε η κατάρτιση για την εργασία, που είναι πολύ σημαντική, να παραμείνει σημαντική. Σε πολλές χώρες όμως υπάρχει τεράστια φοβερή συζήτηση για το θέμα αυτό. Ποια θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα της γενικής εκπαίδευσης, λόγω χάρη στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ή της ε, γυμνασιακής επαγγελματικής κατάρτισης. Τεχνική εκπαίδευση δηλαδή. Σε κάποια κατημέλη αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί υπάρχουν διοικητικοί φραγμοί ω προ τον αριθμό λόγω χάρη των μαθητών. Για την επαγγελματική κατάρτιση των ε, ανηλίκων, των μαθητών δηλαδή. Πολλά κράτη όμως δεν μπορούν να το εφαρμόσουν αυτό. Πολλοί θέλουν να σπουδάσουν ε, οι νέοι σε πανεπιστήμια για να γεμίσουν τα όρια, τα, τις θέσεις της αγοράς ε, εργασίας. Εδώ όμως περιορίζουμε την ελεύθερη επιλογή των νέων. Αυτή είναι μια τάση ε, που ισχύει σε πολλές χώρες. Δεν θα τις κατονομάσω, αλλά αντί να επιλέξουν το σωστό προσανατολισμό στην εκπαίδευση και την το εκπαιδευτικό σύστημα. Ίσως θα έπρεπε εμείς να προβλέψουμε ένα σύστημα παρακολούθησης για να δούμε πώς τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης επηρεάζουν την αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό αυτό για να έχουμε ορθές ε, ποιοτικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο σχόλιο για τον οργανισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Μιλάτε για τη συνεργασία με την Ουκρανία. Θα θέλατε να ε, μειωθεί ο αριθμός των πανεπιστημίων ε, της ανώτατης εκπαίδευσης υπέρ της ε, τεχνικής ανώτερης εκπαίδευσης. Ναι, στην Ουκρανία 70% των πανεπιστημίων παράσχουν σπουδές που δεν ικανοποιούν ιδιαίτερα τους φοιτητές μέχρι την ηλικία των 21-22 και η ποιότητα δεν είναι επαρκής. Είναι λοιπόν άκρος σημαντικό να αναλάβει δράση εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την Ουκρανική κυβέρνηση στις προσπαθίες της. Ευχαριστούμε κυρία Κούνεβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι η Κωνσταντίνα Κούνεβα. Θέλω να ρωτήσω τους εκπρόσωπους των οργανισμών που είναι σήμερα κοντά μας και ιδιαίτερα τον εκπρόσωπο του Eurofound αν τους έχει απασχολήσει το ζήτημα των αυτοπασχολούμενων που σε ορισμένες πτυχές του έχει αρχίσει να γίνεται ένα καλυμμένα παράνομο φαινόμενο. Δεν αναφέρομαι στους εργαζόμενους που είναι αυτοαπασχολούμενοι από πραγματική τους επιλογή. Αναφέρομαι στους εργαζόμενους που απολούνται από τους εργοδότες τους, οι οποίοι στη συνέχεια τους προσλαμβάνουν ως αυτοαπασχολούμενους. Είτε στους εργοδότες που προτείνουν επευθεία συνεργασία σε κάποιον με τον οποίο προτιμούν να συνεργάζονται αντιμετωπίζοντας τον ως αυτοαποσχολούμενο, ενώ στην ουσία έχουν μαζί τους σχέση εργασίας. Έχετε σχετικά στοιχεία. Σας απασχολεί το σοβαρό αυτό ζήτημα. ή αν σκέφτεστε να κάνετε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας και ως συνήθως πρέπει να απαντήσουν οι οργανισμοί σε τόσο πολλές ερωτήσεις. Όσοι βρίσκονται ακόμα εδώ ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Θα μπορούσα να δώσω το λόγο για δύο λεπτά στον καθένα αλλά έχουμε ακόμη δύο άτομα που θέλουν να κάνουν ερωτήσει. Ίσως να ξανάρθετε και ε, να μας ή να μας απαντήσετε γραπτός. Θα βρεθεί τρόπος να πάρουμε τις απαντήσεις μας. try. Uh, we have translators uh, uh, um, Όχι, έχουμε διερμηνία. Περισσότεροι. Ο κύριος Πυρίνσκι, αν μπορείτε να είστε σύντομος. Κυρία Πρόεδρε, εκτιμώ αυτή την ευκαιρία να έχουμε διάλογο με τους τέσσερις οργανισμούς Είναι Η ερώτηση είναι αυτό που θα θέσω και είναι η πρόταση. έχει να κάνει με το επενδυτικό πρόγραμμα του Προέδρου Γιούνκερ και το πώς θα γίνει λειτουργικό. Η αίσθησή μου είναι, Πρόεδρε, ότι η τεχνογνωσία των οργανισμών αυτών αποδείχθηκε για άλλη μια φορά σε αυτή την συνεδρίαση και ο αντίκτυπος στην εργασία, στην κατάρτιση, σε όλο το πλαίσιο ε, της απασχόλησης θα πρέπει να αξιοποιηθεί πολύ εντατικότερα. Εν ώψη της επεξεργασίας των κριτηρίων για να επιλέξουμε τα επενδυτικά προγράμματα. Να σας θυμίσω τις πληροφορίες που είχαμε το πρωί. Όταν μιλήσαμε για, την, ε, για το συνδυασμό των κριτηρίων με γεωγραφικά και τομεακά ε, με γεωγραφικές και τομαϊκές παραμέτρους. πιστεύω ότι μεταξύ των εμπειρογνωμόνων που θα συνδράμουν το Διευθυντική Επιτροπή του Ταμείου θα πρέπει να συμμετέχουν και οι δικοί σαν αυτούς που ακούσαμε μόλις τώρα, ώστε να καθοδηγήσουν την επιλογή ε, σε επενδύσεις που δεν θα επιλέγουν μόνο βάση του κερδοφορίας του στην αγορά. Βεβαίω να υπάρχει οικονομική βιωσιμότητα, όμω αν θέλουμε 18% επιστροφέ, απόδοση δηλαδή των επενδύσεων, σε σύντομο ε, διάστημα. Δεν ξέρω αν τελικά το πρόγραμμα θα κάνει τις αλλαγές που θέλουμε στην Ευρώπη. Είναι εντελώ προφανές. Το τι εννοεί η Ευρώπη. Οι οργανισμοί λοιπόν αυτοί μπορούν να μας δώσουν μια εικόνα για το πώς θα εντοπίσουμε οικονομικώς ενδιαφέροντα προγράμματα αλλά για να υπάρχει και όσο το δυνατόν περισσότερη απασχόληση και δραστηριότητε απασχόληση και παβώ διότι τελειώνει ο χρόνο μου, αλλά ελπίζω ότι έγινα σαφή. Ευχαριστούμε κύριε Πυρίνσκι. Η κυρία Ζανόκα. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Απλώς να συνεχίσω στο θέμα του συντονισμού για το σχεδιασμό της έρευνας. Ήμουν εισηγήτρια στην ε, ε, δουλειά της Eurostat για το πώς οργανώνονται οι διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Το ερώτημά μου και πρότασή μου είναι ότι ελπίζω νέο συντονισμός μεταξύ των ε, οργανισμών να επεκταθεί και στο έργο του Eurostat με τις ad hoc μελέτες που αφορούν την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις για να μην ε, επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Να υπάρξει συντονισμός και πρόσθετη αξία στα προγράμματα. Εξ όσων γνωρίζω υπάρχει σχετική επικάλυψη και ένα πρόβλημα συντονισμού στην έρευνα, στις μελέτες, ιδίως σε ό,τι αφορά τον ΩΣΑ και το Eurofund. Σας εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστούμε να συνεχίσουμε. Αν ήθελε κανείς να κάνει μια ερώτηση, τώρα είναι η στιγμή. Παρακαλώ, ε, θέλατε, θέλατε. Με ένα πιο γενικό θέμα θέλω να θέσω, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των οργανισμών για τις παρουσιάσεις τους. Θέλω να πω και κάτι γενικό. Παρόλο που είναι καλό να έχουμε διμερείς σχέσεις για πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πολλά στοιχεία μας ανέφεραν. Κατά τη γνώμη μου όμως υπάρχει ένα στοιχείο που θα έπρεπε να είναι κοινό και θα έπρεπε να είναι αυτό που μας ενώνει και αυτό είναι ότι όλα συνδέονται με τα παραγωγικά μοντέλα και με τις εργασιακές σχέσεις που έχουμε στις διάφορες χώρες. Και είναι περίπλοκο πώς να μιλήσουμε για κατάρτιση, για κοινωνικό διάλογο, για εκπαίδευση, για ε, μετακίνηση των νέων, για την γύρανση του πληθυσμού από κοινού, όταν η πραγματικότητα στις χώρες του Νότου ή στις χώρες ε, στο ανατολικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο διαφορετική. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν καθόλου βιομηχανικό ιστό και δεν πρόκειται να δημιουργηθεί με το επενδυτικό πακέτο Juncker. Εκεί δεν ε, πρόκειται να υπάρξει καινοτομία βιομηχανή, θα χάσουν θέσεις απασχόλησης. Οι νέοι σπρώχνονται προς άλλες χώρες. Οπότε η κινητικότητα τελικά είναι αναγκαστική, δεν είναι σε θελοντική βάση. Δεν υπάρχει κοινωνικός διάλογος επίσης σε πολλές χώρες εξαιτία των εργασιακών μεταρρυθμίσεων. Οπότε αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι ή που θα συντονιστούμε με το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα, με τους στόχους του 2020 και τα λοιπά την καινοτομία ή αλλιώς πολύ ωραία είναι αυτά που μας είπατε αλλά στην πραγματικότητα δεν θα έχουν κανέναν αντίκτυπο ή ελάχιστο αν δεν προχωρήσουμε πιο συντονισμένα στις βασικές μας πολιτικές που είναι η αγορά εργασία, τα παραγωγικά μας μοντέλα κλπ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Φυσικά και επικεντρωνόμαστε όπως καταλάβατε στο επενδυτικό πακέτο. Επίσης σε θέματα μετανάστευσης και αυτά μας απασχολούν. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αν ο καθένας από σας τώρα, σύντομα, θα μπορούσε να μας δώσει κάποιες απόψεις. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, έτσι φαντάζομαι, δεν γίνεται. Αλλά βλέπετε τι είναι αυτό που μας καίει. Οπότε θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Καγέχα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι ερωτήσεις που ακούστηκαν. Στην εισαγωγή μου είπα ξεκάθαρα ότι οι ευρωπαϊκοί αυτοί οργανισμοί όλοι, όχι μόνο εμείς, φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Με αυτό ξεκίνησα και πηγαίνουμε πιο κοντά στους Ευρωπαίους, είτε με τις έρευνές μας, είτε με την ανάλυση πολιτικής. Στόχος μας είναι όλα αυτά να στηρίξουν τελικά τις διάφορες πλευρές. Οπότε αυτό που μας ρωτήσατε πριν που λέτε πού βλέπετε εσείς τη δύναμή σας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η απάντηση είναι ότι συμμετέχουν όλοι οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, οι μαθητές, οι ε, κυβερνήσεις, για να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Όσον αφορά τώρα την εγγύηση για την νεολαία, όλα αυτά πρέπει να βγουν στο κοινωνικό πλαίσιο που ζει ο καθένας. Πολλές φορές το copy-paste, αν αντιγράφουμε δηλαδή και εφαρμόζουμε την ίδια λύση παντού, αυτό δεν λειτουργεί. Γι' αυτό και ως οργανισμός θέλουμε να είμαστε πιο κοντά στις χώρες μέλη, και όχι μόνο στους τεχνικούς, αλλά και στους νέους, στους πολίτες της κάθε χώρας για να καταλάβουμε ποιες είναι δικές τους ανάγκες, ποια είναι τα οράματά τους, ποιες είναι οι ευκαιρίες που αποζητούν. Αυτό που είπαμε εμείς, ε, the roots and the roots, δηλαδή από τις ρίζες στους νέους δρόμους, είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Υπάρχουν όντως μακροχρόνια άνεργοι και έχουμε μελέτες. Αυτό όπως επίσης και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ανεργία έχοντας χαμηλά προσόντα. Και έχουμε κάνει συστάσεις. Το άλλο βέβαια θέμα είναι πώς μέσα στο σύστημα οι συστάσεις αυτές θα λειτουργήσουν για τους πολίτες. Μία από τις φετινές μας πρωτοβουλίες είναι να έχουμε κάποια φόρα για τις χώρες μέλη όπου συζητάμε συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή με σημείο κίνηση στις ευρωπαϊκές πολιτικές προσπαθούμε να τις θέσουμε στα διαφορετικά εθνικά πλαίσια, στις διάφορες χώρες μέλη. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία, πιστεύω, που θα έπρεπε να οδηγήσει στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών, κάτι που είναι ο βασικός μας στόχος για την περίοδο 2016-2020. Ο βασικός μας στόχος δηλαδή είναι να δούμε πώς εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Πολιτικές που θα βοηθήσουν τους ε, μαθητές, τους εκπαιδευόμενους να προχωρήσουν. Γιατί τι λέμε ότι θέλουμε, απασχόληση, μισθούς, με ποιότητα ζωής. Πώς θα το προσεγγίσουμε αυτό, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και για να το κάνουμε αυτό ερχόμαστε σε επαφή όχι μόνο με τους τεχνικούς αλλά και με τους πολίτες. Και εσείς είσαστε το σωστό φόρουμ όπου πρέπει να περάσουμε αυτό το μήνυμα και εσείς με τη σειρά σας πιο πέρα. Δηλαδή από τα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας, εκεί που βρίσκονται οι μαθητές, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις. Αυτή θα είναι μια βασική μας προτεραιότητα για την περίοδο 2016 με 2020. σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Μενέντεθ Βαλντές τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω με κάτι πολύ συγκεκριμένο που ρωτήσατε στην Ευρωβουλευτή από την Ελλάδα για τους αυτοπασχολούμενους. Έχουμε μία έρευνα και έκθεση που λέμε ότι δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Αυτή την έκθεση μπορούμε να σας την δώσουμε και έχουμε συμπεριλάβει και άλλα ζητήματα και έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα φέτος ακριβώς για την ψεύτο αυτοπασχολούμενη εργασία. Αντιμετωπίζουμε διάφορες συμβατικές μορφές που δείχνουν ένα νόμιμες χωρίς όμως να είναι ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε, προσπαθούμε λοιπόν λοιπόν να μπούμε και στην πλατφόρμα για την αδήλωτη εργασία που έχει φτιαχτεί. Στην κυρία Στάινβερκ θέλω να πω ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ φυσικά να πω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά η ποιότητα των θέσεων απασχόλησης φυσικά είναι κάτι που μετράμε. Πολλές από τις ερωτήσεις που έχουμε στην έρευνά μας έχουν να κάνουν με αυτό. Δεν μπορώ τώρα να σας τα πω, αλλά αν θέλετε διμερώς μπορώ να σας τα εξηγήσω. Παρακολουθούμε τις τάσεις, τι θέσεις απασχόλησης έχουμε στην Ευρώπη σήμερα. Και αυτό έχει να κάνει και με την ερώτησή σας για το τι αγορές εργασίας φτιάχνουμε. Έχουμε διάφορα προγράμματα. Εξετάζουμε τις ε, πολιτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν λειτουργήσει. Είναι δύσκολο βέβαια να δούμε μια συνολική μεταρρύθμιση και να την αξιολογήσουμε κοιτάμε τα επιμέρους μέτρα και προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία και αξιολόγηση, κάτι το οποίο βέβαια δεν βρίσκουμε πολύ εύκολα στην Ευρώπη. Ευελιξία. Βέβαια θέλουμε και μερικές φορές είναι πετυχημένη αυτή, αλλά πρέπει να δούμε τι θέσεις απασχόλησης δημιουργούμε και κατά πόσο αυτές είναι βιώσιμες, κατά πόσο είναι θέσεις δηλαδή που θα κρατήσουν στο χρόνο. Γιατί και εδώ είναι θέμα επιλογής που θα κάνουμε για να έχουμε απασχόληση βιώσιμη που να αντέχει στον χρόνο. Αναφερθήκατε στον κοινωνικό διάλογο επίσης. Υπάρχουν παραδείγματα. Κοινωνικό διάλογο έτσι καλώς έχουν ακόμα και χώρες που υπέφεραν πιο πολύ. Έχουμε τις επιπτώσεις βέβαια της κρίσης τις, στις χώρες ιδίως που βρίσκονται σε πρόγραμμα και ξέρουμε ότι ο συντονισμός και η διάρθρωση μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων είναι ζωτική σημασία σε κάθε χώρα μέλος. Οπότε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν πάμε από το εθνικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τη νέα οικονομική διακυβέρνηση, πρέπει να δούμε πώς θα έχει η διάρθρωση αυτή του εθνικού κοινωνικού διαλόγου. Και θα τελειώσω με την κυρία Λόπεθ. Στα ισπανικά θα τις απαντήσω, μια που είναι η μητρική μου γλώσσα τα ισπανικά. Παλώμα, για αυτό που ρώτησες. Αυτά που λες έχουν να κάνουν με τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουν οι πολιτικοί, αυτοί που αποφασίζουν. Εμείς οι οργανισμοί στοιχεία προσφέρουμε, πληροφορίες και διευκολύνουμε το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Αλλά συμφωνούμε με αυτά που είπες. Έχουμε ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή για τις διαστάσεις των ε, συστημάτων εργασιακών σχέσεων σε κάθε χώρα. Δεν λέω ότι πρόκειται για ένα πίνακα επιδόσεων, αλλά πάντως συμπεριλαμβάνουμε διάφορα στοιχεία για το τι ισχύει από αυτού στην κάθε χώρα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Σέντλατσεκ τώρα. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω κι εγώ στα γερμανικά στην κυρία Στάινρικ. Για το Refit, όχι, δεν συμμετείχαμε γιατί τότε το έγγραφο θα είχε λάβει άλλη μορφή. Ο στόχος βέβαια ήταν η απλοποίηση, η απογραφειοκρατικοποίηση, ιδίως ό,τι αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς βέβαια προσυπογράφουμε αμέσως και γι' αυτό φτιάξαμε και αυτό το όιρα που σας εξήγησα προηγουμένως για να βοηθήσει τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όμως βέβαια προσοχή διότι αυτό μαθαίνουμε από την εμπειρία μας σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις συχνά το ποσοστό των ε, ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών είναι πολύ υψηλότερο. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει νομική βάση, βεβαίω αυτή πρέπει να ισχύει ισοδίκαια για όλου, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι βεβαίω οι μεγάλε επιχειρήσει έχουν και συστήματα ανάπτυξη που βοηθούν στην αποφυγή ατυχημάτων κλπ. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν αλλαγή τη νομοθεσία. Αυτό που χρειάζεται είναι ενισχυμένη υποστήριξη των μικρών και των μικροεπιχειρήσεων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τώρα, για το σύστημα OIRO που σα εξηγήσαμε προηγουμένω, έχουμε και άλλα ηλεκτρονικά εργαλεία στο πρόγραμμά μας Αυτά που δημιουργούμε δηλαδή είναι μια συλλογή, αξιολόγηση και διανομή, ή κατανομή των ηλεκτρονικών εργαλείων για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εμπειρογνώμονες των χωρών μελών για να αναπτύσσουμε τα συστήματα αυτά έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Δεν θα αναπτύσσουμε τα tools αυτά εμείς ψάχνουμε να βρούμε που είναι τα καλύτερα. Έχουμε φτιάξει τώρα και μια ειδική ιστοσελίδα. Είναι ένα έργο το οποίο συνεχίζεται και ασφαλώς βοηθεί πολύ τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για την Ευρωστάτ στην δραστηριότητά μας όταν πρόκειται για παράδειγμα για ε, την ε, επιθεώρηση ΕΣΕΝ ή για τις επαγγελματικές ασθένειες πάντοτε πρώτα ερχόμαστε σε επαφή με την Ευρωστάτ. Δεν υπάρχουν δηλαδή επικαλύψεις δεδομένων ή ε, αναλύσεων. Έχουμε συνεργάτες που έχουν αναλάβει ακριβώς αυτή την επαφή με την Ευρωστάτ για να αποφύγουμε επικαλύψεις. Τώρα, για το σχέδιο επενδύσεων, η συζήτηση βεβαίω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Κάτι που με απασχολεί και το λέω ως ε, παράδειγμα μόνο, ο οργανισμός μας, η EU OSA, έχει ένα δίκτυο και στις 28 χώρες μέλη. Εμείς συνεργαζόμαστε με το δίκτυο τρεις φορές τον χρόνο για την ασφάλεια και προστασία των εργαζόμενων. Είμαστε λοιπόν πολύ κοντά στην βάση και εάν θέλουμε να δούμε κάτι σχετικά με το σχέδιο επενδύσεων που θα μπορούσε να κάνει στην περίπτωση αυτή, θα ήταν να συνεργαστεί με το δίκτυο αυτό και να δούμε πού μπορεί να βοηθήσει κάποια υποστήριξη, πού μπορεί να είναι πραγματικά αποδοτική, να δοθεί δηλαδή από το σχέδιο επενδύσεων κάποια υποστήριξη. Αυτό που κάνουμε πάντα βεβαίως είναι σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και το δίκτυό μας στην κάθε χώρα μέλος. Αυτό αποτελεί μεγάλο κέρδος για όλους, διότι όλοι συμμετέχουν και βεβαίως εμείς αντλούμε ιδέες από όλες αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ. Η κυρία Σέρμπαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που μας ε, έδωσαν με τις ερωτήσεις τους κάποιους προσανατολισμούς. Να είμαι πολύ σύντομη, δεν μπορώ να επαναλάβω όσα υπόθηκαν. Απλώς νομίζω ε, αναφέρθηκε και ευχαριστώ την κυρία Στάινμπρουκ που, Στάινρουκ που το είπε, που ευχαρίστησε όλους μας για τη δουλειά μας, το ίδιο και για τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τους συναδέλφους που κάθονται πίσω, είναι μια συλλογική προσπάθεια ότι κάνουμε και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, προεδρεύει στο Διοικητικό μα Συμβούλιο. Ευχαριστούμε για όσα πετύχαμε στο, το 2014. Νομίζω ο κοινωνικό διάλογο, τα κοινωνικά κεφάλαια που ανέφερα στην αρχή, είναι μάλλον το θέμα, θα, είναι, μπορούσε να είναι ένα θέμα του ερχόμενου σεμιναρίου των τεσσάρων οργανισμών. Ε, όχι γιατί έχουμε εργαστεί μόνο από αυτού, αλλά γιατί είναι ζωτική σημασία. Έχουμε πολλά αποδεικτικά στοιχεία από όσα κάνουμε με τι χώρε εταίρους που ε, τη στήριξη και την ε, συνδρομή την ε, έχουν αξιοποιήσει καλύτερα εκεί που λειτουργεί και η διακυβέρνηση. Η διακυβέρνηση πρέπει να συνδυάζει εργοδότε, εργοζομένου, την κοινωνία των πολιτών και τι τοπικέ αρχέ. Νομίζω ότι μπορούμε ω οργανισμό να δείξουμε πώς, πώς μπορούμε να εμπνευστούμε από την Ευρώπη και τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τα σε συμβούλια σε όλες τις χώρες, φροντίζοντας να συμμετέχουν στις κρατικές πολιτικές. Εάν λοιπόν θεωρείτε ότι αυτό είναι ε, ενδιαφέρον, ευχαρίστως με τη στήριξή σας να βρούμε μια ημερομηνία και να προχωρήσουμε για μια τέτοια συζήτηση, για το πόσο ο κοινωνικός διάλογος ε, και οι υπηρεσίες μπορούν να εμπνεύσουν ε, τις δημόσιες πολιτικές, όποιες και είναι τομέας δράσης. Και να ευχαριστήσω, παρόλο που λείπει, την, ε, την βουλευτή από την Τσεχία, η οποία είπε ότι οι κρατικές πολιτικές, εάν δεν έχουν κοινωνικό όφελος, δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Διότι μπορούμε να έχουμε 2.000 δείκτες, αλλά αν οι πολίτες δεν έχουν την αίσθηση ότι οι πολιτικές τους εξυπηρετούν σε κάτι, δεν χρησιμεύει σε τίποτα όλο αυτό. Έχουμε πόδινες εμπειρίες από τα διδάγματα του παρελθόντος. Στην Τινησία δεν ξεχάσαμε τι έγινε με την γραφική άνοιξη που... Ε, ξεκίνησε με κοινωνικά κινήματα ε, πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης που είχαν την ένδειξη ότι για την ανάπτυξη της χώρας τους δεν θα είχαν κανένα μέλλον έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί τα πράγματα. Καμία προοπτική για τη ζωή τους. Γι' αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλες τις χώρες και να δούμε ποιο είναι ε, το σημείο που μπορούμε να συνδυάσουμε τις προσδοκίες τους με τις ε, φιλοδοξίες που έχουν για τη χώρα τους. Και αυτό με φέρνει στη μετανάστευση, διότι όπως είπα η μετανάστευση είναι κάτι που έχει ξεφύγει του έλεγχου μας. Ε, δεν ε, μπορώ να επηρεάσω όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαι απλώς από, το, από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ε, αλλά αν μπορεί η φωνή μου να ακουστεί, ε, παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι στις χώρες προέλευσης πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, όχι μόνο από τις κυβερνήσεις, αλλά και από τους εργοδότες και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και η επιστροφή των ψηφοφόρων η επιστροφή μάλλον των μεταναστών πρέπει να γίνει προς τα εκεί. Μπορούμε πάντως να παρουσιάσουμε τα πορίσματα των μελετών μας και να στηρίξουμε έτσι τις εργασίες σας. Αυτά από την πλευρά μου σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις σας και τις απαντήσεις και αυτές τις τόσο τεκμηριωμένες παρεμβάσεις. προς τους οργανισμούς να πω αυτό που είχα πει και την περασμένη φορά νομίζω που είσαστε εδώ. Καλώς μας ήρθατε. Κυρίσω τη λήξη της συνεδρίασης, επόμενη συνεδρίαση στις 3, ε, 3 Φεβρουαρίου και στις 26 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ, γεια σας.